Dear colleagues, please take your seats. Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μετρήσω αντίστροφα στα ελληνικά από το 10 στο 1 και μετά θα αρχίσω. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2010 η διάσκεψη των προέδρων ενέκρινε σύσταση για την παράταση της θητείας της ειδικής επιτροπής για την χρηματοπιστωτική οικονομική και κοινωνική κρίση η οποία κανονικά λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2010 έως την 31η Ιουλίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 184. Υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά αυτή τη σύσταση. Δεν υπάρχουν. Η σύσταση εγκρίνεται. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής για τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση παρατείνεται δια της παρούσης ως την 31η Ιουλίου 2011. Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία επ' της έκθεσης της κυρίας Χάουταλα σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συγγήτρια η κυρία Χάουταλα θα ήθελα να προτείνει δύο προφορικές τροπολογίες σε αυτήν την έκθεση. Κυρία Χάουταλα, έχετε το λόγο. Ε, President, Πρόεδρε, φαίνεται να είναι ευρία η συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων για δύο προφορικές τροπολογίες στην έκθεση αυτή και η μία συνδυάζει την παράγραφο 6 και 22 και θέματα εμπορίου να μπουν στην ίδια παράγραφο και η δεύτερη αφορά μία αναδιατύπωση της παραγράφου 19 ε, για τη λογοδοσία και θέλω να εγκριθούν, νομίζω μπορούν. Δύο τροπολογικές τροπολογίες. Όχι. Άρα με μόνη ψήφο συμπεριλαμβανομένων των προφορικών τροπολογιών για την έκθεση Χάουταλα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Κλίντς σχετικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Ψηφίζουμε το μπλοκ νούμερο 1 Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το μπλοκ 2 καταπίπτει. Ε, η ψήφος επί της τροποποιημένης πρότασης. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με ονομαστική κλίση η ψήφος επί του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κλίντς. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία τη έκθεση του κυρίου Ρωμέβα Ιρουέντα σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλλιευμάτων για τον τόνο. Τούνους θύμνους για όσους ενδιαφέρονται. Μπλοκ 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το μπλοκ 2 καταπίπτει. Ψήφος επί της τροποποιημένης πρότασης. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με ονομαστική κλίση το ψήφισμα. Άρκετη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται Συγχαρητήρια στον κύριο Ρωμέβα Ιρουέτα. Η ημερήσια διάταξη προβλέψει ψηφοφορία της του κυρίου Κοέλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σέγγεν όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψήφος επί της τροποποιημένης πρότασης. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Με ονομαστική κλίση το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κουέλιο. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία τη πρώτη ψηφίσματο τη Επιτροπή Οικονομική και Νομισματική Πολιτική σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και τι ενισχυμένε ελεκτικέ εξουσίε τη Επιτροπή Eurostat. Μία και μοναδική ψήφο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία επ' της έκθεσης του κυρίου Ρωμέβα Ιρουέντα σχετικά με την διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η παράγραφος 1 με ονομαστική κλίση άρκετη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η παράγραφος 3 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. I don't see it here. Is With call vote. Πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Με ονομαστική τα είπα και τα δύο. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρι... Ε, απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σε δύο μέρη Oh, we're not going to have this thing again, are we? Okay. Πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε. Let's check. Ωραία, έλεγχος. Τροπολογία 1. Α, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Παράγραφος 13. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Πάλι. Again. Παράγραφος 13. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Με ονομαστική κλίση. άρκετη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20 σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 21. Σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 28. Σε τρία μέρη και τα τρία με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 31 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 40 σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η τελική ψήφος με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Ρωμέβα Ιρουέντα. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Φουικοϊρέδο σχετικά με την αξιολόγηση του χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον. Κυρία Λούλιν, έχετε ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Θα ήθελα στο άρθρο 175β να αναφερθώ του κανονισμού και εξ ονόματος της ομάδας μου να ζητήσω αναπομπή της έκθεσης αυτής ε, στην Επιτροπή. Συγκρίναμε μεθοδικά την έκθεση Ρομέβα που μόλις ψηφίσαμε την έκθεση Φιγκερέδο και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ταυτόσιμες ακριβώς παράγραφοι για στις δύο εκθέσεις. Αιτιολογικές σκέψεις, το διατακτικό, άρθρα, ακριβώς τα ίδια εντάξει, όχι επιλέξει, αλλά ε, το νόημα είναι το ίδιο. Και η έκθεση αυτή τι κάνει. Σε μεγάλο βαθμό αναπαράγει αυτά που ήδη έλεγε η έκθεση Ταραμπέλα παλαιότερα για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Και την ψηφίσαμε εδώ το Φλεβάρι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι εισηγητές που δεν έχουν έμπνευση και ε, είναι ε, υπεύθυνοι για αυτή την αντιγραφή αλλά το κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να γίνει περίγελος. αυτό θα πρέπει να αναπέμψουμε την Επιτροπή, την έκθεση γνώμη στην Επιτροπή. Επιπλέον και εκτός θέματος, ξέρετε. Κύριε Λούλινγκ, ξέρετε πως δεν είναι ώρα για ομιλίες και για χορεύσεις. Έχετε μεγάλη εμπειρία. Δεν καταλαβαίνω γιατί στην Επιτροπή Γυναικών συνεχίζει, κυρία Λούλινγκ. Η έκθεση αυτή έγινε αποδεκτή. Δεν είναι καλή νομοθετική δουλειά. Να πάει ξανά πίσω στο εργοστάσιο. Okay. I will take one... Συνάδελφοι, θα ακούσουμε έναν υπέρ και έναν κατά. Ποιος θέλει να μιλήσει υπέρ του αιτήματος της κυρίας Λούλινγκ. Who Κανείς φαντάζομαι καλύπτεστε από τα όσα είπε η κυρία Λούλινγκ. Κατά ποιος θέλει να μιλήσει. Ε, Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Φιγερέδο, η κυρία Λούλινγκ Η κυρία Λούλινγκ και το ΕΛΚ γνωρίζουν ότι έγινε μια πολύ έντονη συζήτηση για αυτή την έκθεση και ότι συγκέντρωσε τις συμβολές ε, βουλευτών από όλα τα κόμματα ή σχεδόν όλα τα κόμματα και ότι υπήρξε μια ψηφοφορία σαφώς πλειοψηφική στην Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Η πλειοψηφία υπερψήφισε. Μόνο δύο ψήφοι κατά υπήρξαν. Ήταν η κυρία Λούλινγκ και κάποιος άλλος βουλευτής και καμία, κανείς άλλος. Η πλειοψηφία λοιπόν ήταν υπέρ. Καμιά ομάδα δεν απήγε. Άρα λοιπόν, εντάξει, η δική της γνώμη είναι αυτή, αλλά δεν είναι η γνώμη της πλειοψηφίας στην Επιτροπή. και ε, κανονικά είναι και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου που σκέφτεται το ίδιο. Η ίδια η Επίτροπος, η κυρία Ρέντινγκ, την Τρίτη το βράδυ εκφράστηκε υπερθετικά για αυτή την έκθεση, όπω όλοι γνωρίζουν που συμμετείχαν στη συζήτηση. Θεωρεί πως είναι πολύ χρήσιμε προτάσει για τη νέα στρατηγική που βρίσκεται υπό προετοιμασία για την ισότητα α, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και προτείνω ή να την υπερψηφίσετε την έκθεσή μου. Ωραία λοιπόν. Θα θέσουμε το αίτημα για την ε, παραπομπή στην Επιτροπή σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της παραπομπής στην Επιτροπή. Ποιοι είναι κατά. Okay. Let's check this. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αν έρχεται η ψηφοφορία. The vote Τέλος ψηφοφορίας. So it was rejected. Απορρίπτεται. Okay. The request was rejected. Ωραία, λοιπόν, το αίτημα απορρίπτεται και άρα προχωράμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι... If you don't quiet down... I'm not checking. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Check. Τροπολογία 6. Check. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Is 21. Ε, η α, παράγραφος 21 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Okay, I will check one last time. Εντάξει, τελευταία φορά. Ε, αλλά έχω δίκιο τώρα, ποτέ ξανά δεν θα ελέγξουμε. Συμφωνείτε, εντάξει. Ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 36 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, με συγχωρείτε. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 71 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 72 σε δύο μέρη. Α, με συγχωρείτε. Τροπολογία 1. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 72 σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 73 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 74 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 77. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Recital E σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Recital N. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο μέρος ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται recital AC ποιος θα μου πει πως είναι το AC στα ελληνικά παρακαλώ κανείς is AC in Greek? Doesn't matter for now. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στο Recital S υπάρχει μια προφορική τροπολογία από την κυρία Βερζιά. Κυρία Βερζιά, έχετε το λόγο. Α, την έχει αποσύρει. Thank you very much. I got it. Recital S, νέο ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας οφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Okay, okay. Check, final vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Φιγκορέντο. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της πρώτη απόφασης της διάσκεψης των Προέδρων με θέμα την ίδρυση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Δεν υπάρχουν τροπολογίες, οπότε η πρόταση είναι αυτομάτως αποδεκτή. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με τους μάνετζερ ποδοσφαιριστών στον αθλητισμό. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία των έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με το αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία που έγινε στο Ροστόφ επί του Δον στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2010. Πρώτα ψηφίζουμε στην πρόταση ψηφίσματος των Πρασίνων. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά αποχές απορρίπτεται πηγαίνουμε τώρα στο κοινό ψήφισμα παράγραφος 2 με μια προφορική τροπολογία που προτείνει ο κύριος Σαρουσβόλσκι κύριε Σαρουσβόλσκι έχετε το λόγο Mr. Chairman, uh, I propose that... Uh, Κύριε Πρόεδρε, προτείνω όταν μιλάμε για αυτή τη δεύτερη παράγραφο για εξυγχρονισμό της Ρωσίας να εκφράσουμε την κατανόησή μας ότι δεν μιλά μόνο για οικονομία, τεχνολογία και κοινωνία που θα πρέπει να καλύπτει τόσο την οικονομία και όσο και την κοινωνία. Άρα, Παράγραφος 2 με την τροπολογία την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 με ονομαστική κλίση. τροπολογία 5 με συγχωρείτε. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Υπάρχει και εδώ. Και στην παράγραφο 10 υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Κύριε Σαρουσβόσκη, you have an amendment, I understand. Έχετε προφορική τροπολογία. Mr. on paragraph 10... Κύριε Πρόεδρε, στην παράγραφο 10 και σύμφωνα με τις ε, θέσεις σχεδόν ομόφωνες που ακολουθεί το Κοινοβούλιο μας και στην έκθεση εξωτερικής πολιτικής για την ενέργεια ανέκαθεν αποκλείουμε την ενέργεια από τη χρήση της ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και γι' αυτό προτείνω να προσθέσουμε τα εξής λόγια αποκλείει την χρήση της ενέργειας ως ένα εργαλείο για εξωτερική πολιτική. Όχι. Άρα παράγραφος 10 με την τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12 σε πέντε μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο μέρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται δεύτερο μέρος άρχεται ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. «Άρκετη η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Με ονομαστική κλίση. άρκετη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα η τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επομένως τα ψηφίσματα των υπολείπων ομάδων καταπίπτουν. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία των 7 προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας. Ο κύριος Τάνοκ έχει ζητήσει point of order. Κύριε Τάνοκ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, ως διαμαρτυρία η ομάδα μου δεν θα ψηφίσει για το ψήφισμα θα το, καταψηφι... το καταψηφίσαμε γιατί οι συντονιστέ των φιλελευθέρων που διοργάνωσαν το κοινό ψήφισμα δεν ε, μπήκαν στον κόπο να μα καλέσουν στου διαπραγματεύσει γιατί υπέθεσαν ότι δεν θα υπογράφαμε το κοινό κείμενο. Στα 11 χρόνια που έχω διατελέσει ευρωβουλευτή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, είναι έναντι κάθε σύμβαση και παράδοση του σώματο και επειδή θα ψηφίσουμε έτσι δεν θα έχουμε κάνει την ευκαιρία να ψηφίσουμε για το δικό μας ψήφισμα. Κύριε Τάνοκ, να σας πω ότι τα όσα είπατε ε, τέργεζαν περισσότερο στην, ως επεξήγηση ψήφου στο τέλος της, των ψηφοφοριών, αλλά σας ευχαριστούμε. Ψήφισματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία των έξι προτάσεων ψηφίσματο σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Τροπολογία 8 Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. απορρίπτεται τροπολογία 4 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση Άρκετη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται τελική ψήφος ποιοι είναι υπέρ Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία των έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ο κύριος Κάτσιν έχει μία προφορική... Well, hold on a second. Κύριε Πρόεδρε, στην παράγραφο 9 προτείνουμε προφορική τροπολογία γιατί είναι λάθος η παράγραφος. Τον αφοπλισμό θα θέλαμε ε, να σβήσουμε. Η ε, εξαμερείς δεν είναι κατά ε, των όπλων, είναι της μη χρήσης πυρηνικών, όχι του αφοπλισμού. Καλούμε τη συνέχιση των συνομιλιών και τα λοιπά, όχι για τον αφοπλισμό, για τα πυρηνικά. Take the word disarmament out of the, of the, of the paragraph, of paragraph 9. Υπάρχει αντίρρηση σε αυτή η προφορική τροπολογία. Όχι. Επομένως ψηφίζουμε την παράγραφο 9 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος επί του κοινού ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τροπολογία 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 σε δύο μέρη πρώτο μέρος ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές I Ηλεκτρονικός έλεγχος στην τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. I will check. Άρχεται ο έλεγχος. Πέρας φορείας. Εγκρίνεται. Okay. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία των πέντε προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Παράγραφος 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 26 σε τρία μέρη πρώτο μέρος ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο μέρος ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψήφος ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος της επιτροπής μεταφορών και τουρισμού σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Υπάρχει μόνο μία τροπολογία, η τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψήφος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία των έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τις πλημμύρες στι χώρε της Κεντρικής Ευρώπης. Ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, ε, Σλοβακία και Ουγγαρία. Κύριε Σβόμποντα, έχετε το λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε αυτό να το προσθέσουμε, αλλά αυτές τις μέρες έχουμε τεράστιες πλημμύρες και καταστροφικές στη Γαλλία. Αν μη τι άλλο, δεν ξέρω πώς θα το διατυπώσουμε, αλλά βάλουμε καμιά πρόταση και γι' αυτό. Ότι λυπούμαστε πάρα πολύ ε, και για τα θύματα των πλημμυρών θα ήταν ε, άκομψο και φοβερό να ψηφίσουμε τέτοιο ψήφισμα χωρίς αναφορά στη Γαλλία. How do we deal with take that as an amendment on the paragraph with the wording proposed by Mr. Swoboda. Κύριε θα πάρουμε αυτό το οποίο προτείνεται ως ε, προφορική τροπολογία με τις λέξεις που βασικά προτείνατε. Υπάρχει αντίρρηση σε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Υπέρ της προφορικής τροπολογίας του κ. Τσουφόβοντα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψήφος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Πέρα ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος πέντε πολιτικών ομάδων σχετικά με την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών. Μία ψήφος μόνο, η τελική, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Μιλάνα σχετικά με μια νέα όθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας. Ο κύριος Γκόλνης ζητάει το λόγο. Κύριε Γκόλνης, έχετε το λόγο. 15 δεύτερα, κύριε Πρόεδρε. Στην επιμόρφωση των δικαστών θα πρέπει να τους ενημερώνετε και τα δικαιώματα των βουλευτών Αυθαίρετα μόλις προσέλαβα να με συλλάβουν με περιφρόνηση πλήρη της ε, κοινοβουλευτικής μου ασυλίας και στη Λιόν τους το έθεσα υπόψη. Παρακαλώ σημειώστε το και ζητήστε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου να απαιτήσει από τις γαλλικές αρχές τις εξηγήσει που απαιτούνται. Ευχαριστώ. Έκθεση Μιλάνα. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 29 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές I'll check δεύτερο μέρος electronic check άρχεται η ψηφοφορία πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται Παράγραφος 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 43. Υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Recital I. Υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Recital J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Recital W. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Recital... Recital X. Υπέρ. Who wants a check on recital w? Ποιος θέλει έλεγχο για το W. Ναι, ξέρω ποιος είστε. Έναρξη ψηφοφορίας. Τέλος ψηφοφορίας. Recital, recital, no, they will live, they will live, Mr. Schultz. Θα ζήσουν, θα επιβιώσουν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψήφος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται have a wonderful weekend colleagues Καλώς σας συνάδελφοι λέει ο Πρόεδρος Προχωράμε στις επεξηγήσεις ψήφου Στην έκθεση Χάουταλα Κύριε Πόσελ, θέλετε το λόγο? Κύριε Πρόεδρε, σας εκτιμώ πάρα πολύ και η Προεδρία σας ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτή την ψηφοφορία. Μόνο μία παράκληση έχω προς όλους τους αντιπροέδρους την Πέμπτη το μεσημέρι να μην εύχεστε καλώς